Η δήλωση της Επιτροπής για τα προβλήματα λυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στα πλαίσια της πρόσφατης υπόθεσης αλογίσιου κράτους δεν ε, θα υπάρξουν μπλε κάρτες και δεν θα υπάρξουν ε, παρεμβάσεις ομιλητών. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Μπόρκ. members, in recent weeks I have addressed Είχα πάρει το λόγο πριν από δύο εβδομάδε στην ε, Επιτροπή Γεωργίας αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της 20 και 21 Φεβρουαρίου. Μετά από την αποκάλυψη ποσοτήτων αλογίσιου κρέατος με εσφαλμένη σήμανση ως βόλιο κρέος και βεβαίως με σκοπό να αποφευχθούν ε, παρόμοιες περιπτώσεις στο άμεσο μέλλον. Το σκάνδαλο αυτό σε καμία περίπτωση όμως δεν αναφέρεται σε προβλήματα, κρίση ή σκάνδαλο που αφορά τη δημόσια υγεία. Οι μέχρι τώρα έρευνες που έγιναν όσον αφορά τα θέματα δημόσιας υγείας μας ε, έχουν ε, δώσει κάποια πρώτα συμπεράσματα που μας οδηγούν ε, στην διαπίστωση αυτή, ότι τουλάχιστον δεν υπάρχουν θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, αλλά πρόκειται για μια απατηλή σήμανση. Τα κράτη-μέλη είναι, όπως ξέρετε, αρμόδια για την καθημερινή υλοποίηση, εφαρμογή των κανόνων για τον έλεγχο εάν τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν κάποιο κίνδυνο για την υγεία και βεβαίως υπάρχει και το σύστημα της ε, ταχείας επαγρύπνησης για θέματα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ε, επαγρύπνηση, αυτός ο συναγερμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παρούσα υπόθεση, κυρία Πρόεδρε, αμέσως ενημερώθηκαν όλα τα κράτη-μέλη και το σύστημα αυτό ταχείας ε, επαγρύπνησης και συναγερμού τέθηκε σε ισχύ και λειτουργήσε ικανοποιητικά. Με αυτόν τον τρόπο οι αρχές των κρατών μελών μπόρεσαν να αντιδράσουν και αντέδρασαν έγιναν οι έλεγχοι DNA και την ίδια ώρα είδαμε ότι οι ουσίες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στο αλογίσιο κρέας απουσίαζαν και στις 13 Φεβρουαρίου έγινε μία συνάντηση των εκπροσώπων του των κρατών μελών. Στις 15 είδαμε την ε, πρώτη δήλωση της Μόνιμης Επιτροπής ε, για την αλυσίδα διατροφής και στις 19 Φεβρουαρίου υιοθετήθηκαν τα πρώτα συμπεράσματα και το σχέδιο δράσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι σήμερα Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Στις 15 Απριλίου θα υπάρχουν και τα τελικά συμπεράσματα και μια έκθεση θα υποβληθεί έτσι ώστε με ταχύτατο τρόπο να δείξουμε ότι επιστρέφουμε στην αξιοπιστία. Βεβαίως πριν τα αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα, ό,τι συμπεράσματα υπάρχουν και στοιχεία θα δημοσιεύονται αμέσως. Την ίδια ώρα ξεκίνησε και μία έρευνα στην Europol και πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η διαδικασία λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια έτσι ώστε να επανέλθουμε στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και σε ένα σύστημα αξιόπιστο. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η απάτη σε καμία περίπτωση δεν ε, θέτει σε αμφισβήτηση τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τομέα των τροφίμων. Πρόκειται για μια νομοθεσία και κάθε φορά που προκύπτει ένα σκάνδαλο ή μια κρίση στον τομέα των τροφίμων θα πρέπει να μαθαίνουμε από την εμπειρία. Το σκάνδαλο αυτό με το αλογίσιο κρέας δεν θα πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση και προσπαθούμε σήμερα να βρούμε τρόπους να επανέλθουμε στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και αναλύοντας όλα τα στοιχεία. Η Επιτροπή λοιπόν σήμερα θεωρεί ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τους κανόνες μας, τους ελέγχους σε τρεις τομείς όσον αφορά τις κυρώσεις, όσον αφορά το επίπεδο των ε, ελέγχων και βεβαίως όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων. Οι κυρώσεις και η έλεγχοι αλλά και η υλοποίηση, η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και των κανόνων είναι κάτι που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας, καθώς και το θέμα των κυρώσεων. Η πρόταση η οποία έχει προετοιμαστεί μήνες πριν ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο ενισχύει τους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα τροφίμων και ζητά από τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις όταν υπάρχει παραβίαση στους κανόνες της αλυσίδας τροφίμων. Και βεβαίως εδώ πρόκειται για τους κανόνες οι οποίοι παραβιάζονται και σκοπός μας είναι να δούμε αυτές οι παράνομες δραστηριότητες ε, να οδηγούν σε τέτοιες κυρώσεις που να είναι αποτρεπτικές. Η πρόταση όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων βεβαίως θα πρέπει ακόμα να βελτιωθεί και να περιέχει και τη δυνατότητα από μέλους των κρατών μελών να ζητήσει ενισχυμένους και συντονισμένους ελέγχους για να αποφευθούν οι ελλείψεις και οι αδυναμίες σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων και ειδικοί έλεγχοι, απαιτήσει για ειδικού ελέγχους σε όλη την αλυσίδα, κάτι που ζητάει η Επιτροπή. Ζητά να υπάρχει ένα σχέδιο για τους ελέγχους, τον οποίο θα εφαρμόζουν βεβαίως όλα τα κράτη-μέλη. Όμως, όπως ξέρετε, αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό σήμερα. Τρίτον, όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη και μέλη εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούν καλύτερη σήμανση όσον αφορά την προέλευση των ε, προϊόντων. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση με την παρούσα κρίση, με το παρόν σκάνδαλο, καθότι βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα κράτη-μέλη που θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία έτσι ώστε να ζητήσουμε να υπάρχει υποχρεωτική σήμανση όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων και για ε, προϊόντα τα οποία βρίσκονται μέσα σε ε, παρασκευασμένα τρόφιμα και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα δημοσιευθεί μία έκθεση. Ανέλαβα την υποχρέωση να επιταχύνω τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης, η οποία θα διατίθεται πάρα πολύ σύντομα. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να ασχοληθεί με την σήμαση των κατεργασμένων τροφίμων. Θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη του καταναλωτή για ενημέρωση, την ε, δυνατότητα της υποχρεωτικής αναγραφής προέλευσης και μια ανάλυση κόστους-οφέλους καθώς και την επίπτωση που έχουν αυτά στην εσωτερική αγορά και το διεθνέ εμπόριο. Και όπως σας είπα κύριε Πρόεδρε είμαι απόλυτα ανοιχτό σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα ότι δεν αποτελεί άμεσο αίτιο αυτού του σκανδάλου και σα υπόσχομαι ότι θα αντιδράσω Καταλήλω μετά τη δημοσίευση της έκθεσης. Μολονότι η σήμανση της χώρας προέλευση δεν θα είχε εμποδίσει το να ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο, παρόλα αυτά θα εξετάσω αυτή την έκθεση, θα φροντίσω να δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατόν και θα ενημερώσω για οποιασδήποτε εξελίξεις. Θα ήθελα να τελειώσω αναφέροντας ότι η εμπιστοσύνη του κοινού είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη έννοια. Συνεπώς, θα ζητούσα από τις χώρες μέλη να συνεχίσουν τις έρευνές τους. Καταλήξαμε σε ορισμένα αποτελέσματα και θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι άμεσα θα κυκλοφορήσουν όλες οι πληροφορίες έτσι ώστε να ρυθμιστεί το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατόν. Και πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμή το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών με αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο. Βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικό να διδαχτούμε από τα διδάγματα αυτού του σκανδάλου. Και θα ήθελα να σας πω ότι θα Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην διατροφική αλυσίδα το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα ασφαλείας διατροφικής αλυσίας. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από τις κρίσεις, τις κρίσεις του παρελθόντος και του παρόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας, γιατί το γεγονός ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα στον κόσμο δεν σημαίνει επουδενή ότι θα πρέπει ε, να επιδοθούμε σε μία αυταρέσκεια. Και υπολογίζω πολύ στην υποστήριξη και τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τους βουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Σιμπέρα. Τρία λεπτά παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη με κύριε Επίτροπε. Σημερίζομαι την άποψή σας όταν λέτε ότι έχουμε τα καλύτερα νομικά συστήματα και για τα τρόφιμα μας και τρόφιμα παγκόσμια. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός ότι διαρκώ έχουμε σκάνδαλα για τα τρόφιμα. Και τώρα καταδεικνύεται πάλι με αυτό το σκάνδαλο πόσο μεγάλε είναι οι διαστάσει των προβλημάτων αυτού του τομέα. Και νομίζω δεν θα έπρεπε τώρα να πούμε ότι μικρέ αλλαγέ θα κάνουμε, αλλά πρέπει να ελέγξουμε σε βάθο. Και ελπίζω ότι θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό πράγματι. Να υπάρξουν βελτιώσει αυθεντικέ. Δεν είναι ευφυέ να πούμε τώρα τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για του ελέγχου και εμεί θα κάνουμε μόνο επί των θεμελιωδών αρχών κάποιε προτάσει. Ειδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδιαίτερε ευθύνε εδώ, ώστε σε αυτόν τον τομέα να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πράγματα σωστά. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είχαμε τόσο μεγάλη, ε, ότι χάσαμε την εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Να αποκαταστήσουμε τώρα την εμπιστοσύνη των πολιτών σε εμά θα είναι πολύ δαπανηρό και πολύ δύσκολο εγχείρημα. Τώρα, αυτό που είπατε να διακριβωθούν τα πράγματα. Εδώ υπήρχαν εγκληματικέ κινήσει που έγιναν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν μπορούν όλα αυτά απόλυτα να αποφευθούν. Πρέπει όμω να δούμε ποιο σύστημα ελέγχου μπορούμε να εισαγάγουμε, ώστε να είναι πλέον χωρί κανένα ενδιαφέρον οικονομικά για κάποιου να κάνουν τέτοιε, ε, α το πω έτσι, τέτοιου ελιγμού και τέτοιε εγκληματικέ πράξει. Θα πρέπει να υπολογίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο δαπανηρό θα ήταν να είχαμε ελέγχους δειγματοληπτικούς που θα μπορούσαν στο ένα ή άλλο σημείο να αυξηθούν ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να έχουμε ένα σύστημα ελέγχων πραγματικά αυθεντικά ε, αποτελεσματικό. Καλείται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για να διασφαλιστεί αυτό. Δεύτερον, το ποινικό πλαίσιο στα διάφορα κράτη-μέλη πρέπει να ελεγχθεί. Κάποια κράτη είναι υπερβολικά αυστηρά, άλλα είναι πολύ χαλαρά. Πρέπει και αυτό πάλι να προσαρμοστεί. Πανευρωπαϊκά να ισχύουν οι ίδιες κυρώσεις, οι ίδιες ποινές παντού. Τρίτον, όπως είπαμε, πρέπει διακόπτεται χωρίς μικρόφωνο. Δεν υπάρχει διερμηνία λέτε. Δεν υπάρχει διερμηνία αυτό που λέω. Α, εντάξει, ωραία. Τι να κάνουμε, εντάξει, παρόλα αυτά. Μπορείτε να συνεχίσετε παρακαλώ κύριε Ζέμπερ. Λοιπόν, πολύ καλά. Όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα ελέγχων που θα είναι αποτελεσματικό για τον έλεγχο της ευθύνης. Πρέπει πάλι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών σε εμά. Και στην έκθεση που εκπονεί και θα εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει αυτά τα θεμέλια να διασφαλιστούν. Το αίτημα για την ε, συσκευασία, την ετικετοποίηση στο προϊόν από πού προέρχεται για την προέλευσή του είναι σημαντικό σε σχέση με τα σφαγεία για παράδειγμα, για το κρέας. Είναι πολύ χρήσιμα για τους καταναλωτές για να πάρουν τις αποφάσεις ποια προϊόντα θα αγοράσουν, θα καταναλώσουν. Είναι πάρα πολύ ε, επικίνδυνη η νοοτροπία να είναι κανεί τσιγκούνη ε, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσουμε στα τα πράγματα. Είναι εγκληματικό αυτό. Πρέπει πανευρωπαϊκά να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά. Και αυτό είναι ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δυνατόν ανώτερε ε, προδιαγραφέ για να μπορέσουμε να πείσουμε του πολίτε, του καταναλωτέ όταν αγοράζουν ένα προϊόν ότι ανταποκρίνεται στι απαιτήσει του. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Σίμπερ. Η κυρία Μακέβαν για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, στηρίζω τα περισσότερα από όσα είπατε. Ιδιαίτερα αυτό που ακούσαμε όσον αφορά την επιτάχυνση της μελέτης για την σήμανση σε προϊόντα που περιέχουν κρέας κατεργασμένα. Και την ίδια ώρα ξέρουμε ότι εμείς εδώ πριν από δύο χρόνια ψηφίσαμε αυτή την πρόταση γιατί θέλαμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι επιχειρήσεις όσον αφορά όλη την αλυσίδα κάνοντας μία υπεύθυνη σήμανση για προϊόντα τα οποία ξεπερνούν τα σύνορα. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε σήμερα. Βλέπετε ότι σήμερα οι διαδικασίες, οι αλυσίδες περνούν από τη μία χώρα στην άλλη με πολλούς ενδιάμεσους, πολλούς διαμεσολαβητές και αυτό είναι ένας τρόπος να διαφεύγουν των ελέγχων. Με μεγάλη λοιπόν αυστηρότητα και σοβαρότητα θα κοιτάξουμε την πρόταση και θα πρέπει βεβαίως να δούμε το κόστος. Αλλά είδατε πόσα δαπανήθηκαν τώρα από τις κυβερνήσεις και από τον ε, τομέα των επιχειρήσεων από τη στιγμή που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Θα πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούμε επίσης και το θέμα της ασφάλειας. Πολλοί μου λένε ότι από το 2006, όταν έγιναν οι πρώτες προτάσεις νομοθεσίας και όταν ξεκίνησαν οι πρώτοι έλεγχοι, ιδιαίτερα στις μονάδες κατεργασίας του κρέατος. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δούμε πώς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Πώς γίνονται αυτές οι επιθεωρήσεις. Κάθε τρεις, έξι μήνες όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, αυτό το σκάνδαλο, γινόταν αυτή η έλεγχη κάθε τρεις ή έξι μήνες. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι θα υπάρχει στην πρότασή σας, γιατί στον τύπο, στη Μεγάλη Βρετανία διάβασα, ότι ουσιαστικά θα υπάρχει ένας κανονισμός, νέοι κανονισμοί, για τον τομέα του κρέατος. Κύριε Επίτροπε, θέλουμε εμπιστοσύνη, θέλουμε αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και περιμένουμε πολλά από εσά έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα λάθη του παρελθόντος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέιβις για δύο λεπτά έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα πράγματα, πρώτα πράγματα που έκανα πριν από 14 χρόνια ήταν να κάνω μία συνάντηση για θέματα διατροφικά. Όλοι έδειξαν μεγάλη κατανόηση σε αυτό το θέμα και κλήθησαν οι χώρες μέλη να αναλάβουν δράση. Είπα όμως ότι η Επιτροπή εξαρτάται από τις χώρες μέλη. Δεν έχει κάποια δική της αστυνομική δύναμη για να επιβάλλει τον νόμο. Και στο μυαλό μου έρχονται αυτά που βλέπουμε σε πολλές νομοθεσίες. Αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές. Λέτε ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα σήμαση στον κόσμο. Αλλά βεβαίω ε, οι χώρε μέλη, αν δεν το θέσουν σε πρακτική, δεν ωφελεί σε τίποτα. Επιβάλλονται κυρώσει ε, σε χώρε μέλη. Έχουμε διαδικασίε που εξασφαλίζουν ε, τη συμμόρφωση. Έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση που υιοθετείται. Διαφορετική βέβαια. Και έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι διαφορετικές. Από τη μία πλευρά το κοινό περιμένει την αποτελεσματική εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων σε όλες τις χώρες μέλη. Διαφορετικά δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το πρόβλημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει κοινέ κυρώσει σε όλες τις χώρες μέλη. Αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα για την δική σας υπηρεσία. Αλλά θα πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες συζητήσεις, να γίνουν περισσότερες αναλύσεις του τρόπου με τον οποίο οι χώρες μέλη εφαρμόζουν την νομοθεσία. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την, το όλο πλαίσιο, αλλά και το τρόπο ερμηνείας αν δεν το κάνουμε αυτό, εάν ε, δεν το ε, ε, αφήσουμε να φανεί, τότε δεν θα μπορέσει να υπάρξει εφαρμογή του νόμου και αν το αποτύχουμε, αυτό θα απαξιώσει εντελώς τους νόμους και το αποτέλεσμά μας θα ακυρωθεί. Ευχαριστώ κύριε Ντέιβις. Ο κύριος Σλίτερ, τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και εσάς Επίτροπε Τώρα θα ληφθούν μέτρα ώστε να μπορέσουν νέες προτάσεις ε, να εξεταστούν. Χρειαζόμαστε καλύτερες και πιο αποτρεπτικές ε, κυρώσεις. Πρέπει φυσικά να εξετάσουμε ποια είναι η κατάσταση στα επιμέρους κράτη-μέλη. Τα τελευταία χρόνια τι διαπιστώσαμε. Είδαμε, διαπιστώσαμε ότι κρέατα επί πολλά χρόνια κατεψύχοντο αποθηκευόντουσαν και μετά επανερχόντουσαν στην αγορά προς διάθεση. Και αυτό τώρα ήταν και περίπτωση σκανδάλου που είδαμε τώρα πρόσφατα. Έχουμε σκάνδαλο τώρα με το αλογίσιο κρέας που κατέληξε στο βόηο κρέας ως δίθεν βόηο κρέας και υπάρχει και μια ολόκληρη σειρά προβλημάτων και παραπώνων. Εφόσον έχουμε τέτοιου είδου σκάνδαλα, πρέπει να κινήσουμε και να πούμε, να υποθέσουμε ότι υπάρχει συστημικό πρόβλημα. Στο ίδιο το σύστημα υπάρχουν τέτοιε δυνατότητε ε, νόθευση ε, και απάτη. Πρέπει να είναι ισχυρέ αποτρεπτικέ οι κυρώσει, ε, ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Και έτσι ο κίνδυνο πραγματικά να αποφευθεί, να αποσοβηθεί από εκείνου που θα μπορούσαν κάποτε με αυτά τα μέτρα να ανακαλύψουν καλυφθούν και να τιμωρηθούν. Θα πρέπει λοιπόν στα σφαγεία να υπάρχουν ξεχωριστοί ελεγκτέ, ανεξάρτητοι ελεγκτέ. Να μην μπορούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίε να ελέγχουν εσωτερικά το τι συμβαίνει. Μια και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν κρατικέ αρχέ ή άλλε ανεξάρτητε αρχέ που να κάνουν ελέγχου, έχουν επιληφθεί αυτών των ελέγχων οι επιχειρηματίε. Πρέπει επίσημοι έλεγχοι να γίνονται από τι επίσημε αρχέ. Διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Και η προέλευση, η ε, στην ετικέτα η επισήμανση προέλευσης πάλι να μπορεί να ξέρει κανείς ότι πραγματικά θα είναι αυθεντική μια τέτοια επισήμανση. Να γνωρίζουν οι καταναλωτές ποια είναι η πραγματική προέλευση του προϊόντος που αγοράζουν. Με κρέας για παράδειγμα. Να γνωρίζουν ότι εκεί... Ε, εξετράφει και ε, οδηγήθηκε μετά στην κατανάλωση το κρέας ε, από ε, τις κτηνοτροφικές μονάδες. Θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό για την τροφική αλυσίδα να υπάρξει αυτή η ανείχνευση, η χνηλάτιση, ώστε να υπάρξει η χνηλασία, ώστε να υπάρχει δυνατότητα από το αγρόκτημα, από τη μονάδα εκτροφής μέχρι το πιάτο του καταναλωτή να γνωρίζουμε ποια είναι η πορεία αυτών των προϊόντων. Έτσι, σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει όλα αυτά να ελέγχονται. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Είναι σημαντικά επίσης και για την εσωτερική, ενιαία εσωτερική αγορά. Στην ενιαία αγορά οι αλυσίδες αυτές των προϊόντων είναι όλο και μεγαλύτερες, όλο μακρύτερες. Πρέπει να έχουμε μικρές, μικρής απόστασης αλυσίδες και όχι μεγάλες αλυσίδες, μεγάλης πορείας ενός προϊόντος από τον ε, εκτροφέα στον καταναλωτή. Με μικρότερες τέτοιες αλυσίδε τροφίμων μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όλα πρέπει να γίνουν προ όφελο ε, των καταναλωτών. Να συντμηθούν, να μειωθούν οι αλυσίδε αυτέ ώστε να είναι πιο αποτελεσματική έλεγχη. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Βεβαίως μπορεί να υπάρχει κάτι καλό στην όλη ιστορία. Το καλό της ιστορίας είναι ότι επιστρέψαμε στον παλιό καλό χασάπι της περιοχής ε, εκεί που πηγαίνουν οι άνθρωποι και όταν θέλουν να ξέρουν τι αγοράζουν. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Εγώ είμαι υπέρ της αποτελεσματικής σήμασης Θα πρέπει να πω όμως ότι όταν κάποιος θέλει να διαπράξει μια εγκληματική ενέργεια, δίχως άλλο, μια σήμανση δεν την, δεν θα τον αποτρέψει. Κατά την άποψή μου αυτό συνέβη για δύο λόγους. Η αλυσίδα επεξεργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και από την άλλη ασκείται πίεση από τους λιανέμπορους να μειώσουν τη τιμή και να παράσχουν φτηνό κρέας. Δεν υπάρχει κάτι που ε, να αντιστοιχεί στον όρο φτηνή τροφή. Η τροφή κοστίζει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκολσον. Ο κύριος Άγνιου. Πριν από 13 χρόνια η Βρετανική κυβέρνηση ανόητα επέτρεψε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα νομοθεσίας τροφίμων. Και είδαμε ότι αυτό οδήγησε στη σημερινή κατάσταση και σε μια παντελή έλλειψη των αποφάσεων. Είδατε τα σκάνδαλα που αφορούν το βόλιο κρέας και όσον αφορά την προέλευση και όσο βλέπουμε ότι διευρύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο αριθμός των κρατών αυξάνεται, αυξάνονται και οι περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης. Είδαμε ότι σήμερα το αλογίσιο κρέας, το οποίο παρουσιάστηκε σαν ε, βόλιο κρέας, διαπιστώθηκε μετά από αρκετό καιρό νοθείας και θα πρέπει εδώ να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Είδαμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δυνατότητα ε, αντίδρασης. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Άγνιου. Η κυρία Άντερσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή μίλησε για την νομοθεσία αναφερόμενη στις περιπτώσεις απάτης και φυσικά αυτό ισχύει, υπάρχουν τέτοιε περιπτώσεις. Από την άλλη μεριά εμεί, σαν νομοθέτε, θα πρέπει, όπως είπατε, να έχουμε μία υπεύθυνη αντίδραση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα που εμπεριέχονται στην διατροφική αλυσίδα. Βεβαίω μπορούμε να μιλήσουμε για το σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά και ιδιαίτερα όσον αφορά προϊόντα που περιέχουν κρέας, κατεργασμένα προϊόντα θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι στην χώρα από την οποία περνούν αυτά τα προϊόντα, αλλά και θα πρέπει να ενισχύσουμε και να γίνει πιο αυστηρό το σύστημα για την προέλευση των προϊόντων. Θα πρέπει επίση να λάβουν τι ευθύνε του ε, οι ιδιοκτήτε πολυκαταστημάτων, σούπερ μάρκετ που εμπλέκονται στην διατροφική αλυσίδα. Είδαμε παραδείγματο χάρη ότι προϊόντα που στην Βόρεια Ελλανδία παρουσιάζονται σαν τοπικά προϊόντα θα πρέπει να μπορούν να το αποδείξουν αυτό βάσει μιας ενισχυμένης αντισχεφιμότητας έτσι ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά τέτοια σκάνδαλα στο τομέα των τροφίμων. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στην Ολλανδία έχουμε μια νέα παροιμία, ένα νέο απόφθεγμα δεν λέμε να δώσεις ε, ε, κάτι για να ανταλλάξεις ε, αυτό που έχεις αλλά αλλάζεις με το, βό, το βόδι με ένα άλογο υπάρχουν πολλά προβλήματα εδώ για εκείνους που το ο κρέας το παρουσιάζουν ως ο κρέας αλλά είναι ακόμα χειρότερα όσον αφορά την, την υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις σκανδάλων που δεν έχουν ανακαλυφθεί και πρώτα στα κράτη-μέλη ανακαλύπτονται τα κράτη-μέλη κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά. Τι απορρέει από αυτό. Εμείς ζητάμε εδώ και χρόνια να πάψουν οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν που είναι άχρηστες και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το βόδι από το άλογο. Πρέπει να έχουμε ε, λειτουργούντα συστήματα στα κράτη-μέλη ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα κράτη-μέλη. Δεν θα είμαστε σοβαροί αν δεν πάρουμε σοβαρά την ασφάλεια τροφίμων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόργκ έχει το λόγο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι περισσότεροι ομιλητές εστίασαν τις παρεμβάσεις σε δύο ή τρία σημεία. Πρώτον το θέμα των κυρώσεων. Συμφωνώ ότι παρόλο που η υπάρχουσα νομοθεσία βασίζεται σε οδηγίες και δεν έχουμε κανονισμό, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη για άλλα θέματα όπως το περιβάλλον, με πολύ συγκεκριμένες κυρώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι ε, όταν προετοιμάζουμε τα κείμενα των οδηγιών, στη διατύπωση των οδηγιών. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει σήμερα να δείξουμε ότι το έγκλημα δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτο και δεν αποφέρει κέρδος. Και αυτό είναι κάτι, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Ντέβης, που θα πρέπει να γίνει με τα κράτη-μέλη, καθότι οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων δεν μπορεί παρά να υλοποιηθούν, να εκτελεστούν από τα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη, ένας παραγωγός που συνεχίζει να έχει άδεια ενώ έχει αποδειχθεί ότι είχε εγκληματική δραστηριότητα. Οι οικονομικές λοιπόν κυρώσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν στο επίπεδο των κερδών που απέφερε το έγκλημα. Αν το κέρδος παραβίασης της νομοθεσίας είναι υψηλότερο από την κύρωση που επιβάλλεται, καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστούν επάπειρον αυτές οι παραβιάσεις της νομοθεσίας. Σε καμία περίπτωση βεβαίως ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε η νομοθεσία να μην παραβιάζεται ποτέ. Αλλά θα πρέπει οι κυρώσεις να είναι αποτρεπτικές. Και βεβαίως δεν λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχει νομοθεσία υπάρχουν και παραβιάσεις. Άρα προς προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής και να πω ότι τίποτα δεν θα είναι ποτέ τέλειο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να είναι αποτρεπτικές οι ποινές και οι κυρώσεις και έτσι ώστε το σύστημά μας να είναι αποτελεσματικό, όσο αποτελεσματικό γίνεται. Τώρα, μπορούμε βεβαίως να βελτιώσουμε τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους. Το θέμα διάρθρωσης τώρα αυτών των ελέγχων. Αυτό δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των τροφίμων. Όλη η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τη σήμανση, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει από τον παραγωγό, από τον κτηνοτρόφο στην περίπτωση του κρέατος. Κατόπιν ξεκινάει ένα σύστημα ελέγχου από τις εθνικές αρχές, τις αρχές των κρατών μελών. Και η αρμόδια υπηρεσία στην Ιρλανδία που έκανε τον έλεγχο σε ένα σούπερ μάρκετ για κρέας που επολύτω σαν βόλιο κρέας για χάμπουργκερς και εκεί απεδείχθη για πρώτη φορά η απαλικέ, ε, αποκαλύφθηκε αυτό το σκάνδαλο του αλογίσιου κρέατος που είχε ε, ετικέτα βόλιο κρέατος. Το θέμα λοιπόν είναι το σύστημα των ελέγχων να λειτουργήσει αποτελεσματικά, να υπάρξει έλεγχος των ελεγκτών κατά κάποιο τρόπο και να γίνει έλεγχος των προϊόντων, προϊόντων κρέατος στην προκειμένη περίπτωση και για θέματα ασφάλειας των τροφίμων αλλά και για θέματα σωστής σήμανσης. Και αυτό όχι μόνο για θέματα ασφάλειας, επαναλαμβάνω, αλλά και για την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται στις ετικέτες. Όπως είπε η κυρία Μακέιβιν, είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανεξάρτητες επιθεωρήσεις και έλεγχοι και θα υποβάλουμε μία πρόταση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να διεκπεραιώνουν μη κανονικούς και τακτικούς ελέγχους. Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης, θα σας δώσω λόγους για τους οποίους θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα όσον αφορά την σήμανση για τη χώρα προέλευσης και άλλους τόσους λόγους που έχουν υποβάλει άλλα κράτη-μέλη για, την, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην σήμανση όσον αφορά τη χώρα προέλευσης. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα αυτό είναι περίπλοκο, συνεχίζουμε να το επεξεργαζόμαστε Και το θέμα εδώ του κρέατος ε, που ευεριέχεται σε κατεργασμένα προϊόντα όσον αφορά την προέλευση, την διαδικασία παραγωγής, εμπορίας, διάθεση στην αγορά και βεβαίως επαναλαμβάνω εδώ τα επιχειρήματα των κρατών μελών διαφέρουν και θα προσπαθήσουμε ε, να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα μετά από την εξέταση όλων των επιχειρημάτων. Σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο σκάνδαλο δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα εμπόδια στην εμπορία τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την οθεία, την απάτη και σήμερα βλέπετε τις περιπτώσεις αυτών των προϊόντων που πέρασαν από τη Μεγάλη Βρετανία στην Γαλλία και ήταν παράνομα προϊόντα. Και πρόκειτο για εικονικό ο κρέας. Και βλέπουμε ότι από τη στιγμή που παραβιάζεται ο νόμος σε μία χώρα, οι επιπτώσεις ακριβώς επειδή υπάρχει και λειτουργεί η ενιαία αγορά, είναι άμεσες και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην εξάλληψη του συστήματος Schengen. Χρειάζονται αυστηρότερες κυρώσεις, αποτρεπτικές κυρώσεις και καλύτερη έλεγχη και επιθεωρήσεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε και να πούμε ότι δεν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ευρώπη. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό το τελευταίο <coughs> σκάνδαλο, από αυτήν την κρίση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ε, διατροφική αλυσίδα, να μάθουμε από αυτά τα σκάνδαλα, από αυτές τις κρίσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε κάποιοι έμποροι να κλονίσουν την εμπιστοσύνη και να διαταράξουν τη σωστή λειτουργία της ενέας αγοράς. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα εδώ να σας πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε τέτοιες απατηλές δραστηριότητες να μην ξαναεμφανιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αυτό κλείνει τη συζήτησή μας. Περνάμε τώρα στην ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Έκθεση, ε, κυρία Θόν, έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Η κυρία Τούνεν έχει το λόγο για